Τα πρακτικά της παρουσυνεδρίας θα υποβληθούν για έγκριση στο σώμα στην αρχή της προσεχούς περίοδου συνόδου, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μαζί με τα ψηφίσματα που ε, υιοθετήθηκαν σήμερα. Θα καταθέσω και τα ονόματα των όσων επισημένονται μέσα στα κείμενα. Ολοκληρώνεται έτσι αυτή